μετά από την απόφαση της Επιτροπής ΕΚΟΝ να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις σε διοργανικό επίπεδο βάσει του άρθρου 69 C παράγραφος 1 που ανακοινώθηκε στην έναρξη της Ολομέλειας την 4η 1η Φεβρουαρίου δεν έλαβα αιτήματα για ψηφοφορία, επομένως η Επιτροπή θα μπορέσει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μετά